άλογο, ούτως ώστε αμελητή να εγκριθεί αυτό το τόσο ε, σημαντικό νέο νομοθετικό μέσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα λοιπόν τελειώνει η συζήτηση και αν επιτρέπετε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήθειας διάταξης. Η κατάσταση στο Θιβέτ, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ζήτησε κάποιον λόγο. επί της διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω πως η Ισπανική Προεδρία αποχωρεί. Θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το ότι ούτε η Ισπανική Προεδρία ούτε η είπατε εκπρόσωπος θα είναι παρόντες εδώ και οι θέσεις τους θα είναι άδειες. Έσχος. πρόκειται για κίνηση εσχρή έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνου αιρετού θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά μετά την ε, θέση ενισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Να διαβιβάσετε παρακαλώ στους απόντες το ότι την ημερήσια διάταξη την ορίζει το Κοινοβούλιο και όχι το Συμβούλιο και κάποιος από τους δύο ή η Προεδρία ή η Πατήκουρος οσο επρεπε να είναι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. Με ενημερώνουν πως η Ισπανική Προεδρία ανακοίνωσε πως αναγκαστικά θα αποχωρήσει στις 18 και θα ήθελα όμως τώρα να δώσω τον λόγο πάλι στον κύριο Σευκοβίτη, τον Αντιπρόεδρο, να μας εξηγήσει, να κάνει την δήλωση που έχει να κάνει. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Πρόεδρε, και τους έναν άλλον φάκελο. Τώρα περνάω στον επόμενο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έβαλε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, γιατί νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε και θα πρέπει να ξεκινήσουμε περιγράφοντας το ότι η σχέση μας με την Κίνα είναι πάρα πολύ σημαντική, στρατηγική και είχαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώς επειδή έχουμε μια τέτοια στρατηγική σχέση, κάτι τέτοιο μας επιτρέπει να ασχοληθούμε όλα τα ζητήματα και τα πιο ευαίσθητα. Έχουμε ένα επίπεδο επαφών πολύ υψηλό για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που ασχολούν τους πολίτες μας χωρίς να ε, παραβλέπουμε και τις διαφορές μας. Μία από τις οποίες είναι το Θιβέτ. Είναι προφανές πως οι διαφορές με την Κίνα παραμένουν όσον αφορά το Θιβέτ. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το ότι το Θιβέτ έχει παραμείνει κλειστό για το διεθνή μήνυε διπλωμάτες και ανθρωπιστικές οργανώσεις και δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των Λάμα και των Κινέζικων αρχών. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής, οπότε θα ήθελα να τονίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Θιβέτ. Αλλά πάντα υποστηρίζαμε την ειρηνική συμφιλίωση μέσω του διαλόγου μεταξύ των κινέζικων αρχών και των εκπροσώπων του Δαλάη Λάμα. Διάλογος πρέπει να είναι επικοδομητικός και ουσιαστικός. Να αντιμετωπίζει όλα τα βασικά ζητήματα όπως η διατήρηση του πολιτισμού, της θρησκείας και των παραδόσεων του Θιβέτ, και το ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αυτονομία του Τιβέτ εντό του Κινέζικου Συντάγματο. Επίση ο διάλογο θα πρέπει να δει την συμμετοχή των Θιβετιανών στη λήψη αποφάσεων, γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Θιβέτ είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμεί σταθερά δίνουμε αυτό το μήνυμα στου κινέζου ομολόγου μα και ακούμε προσεκτικά τι απόψει του και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι απόψη ένα πνεύμα αμοιβαία σεβασμό, όμω τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και δικαίως ανισχύει η διεθνής κοινότητα για την κατάσταση στο Θιβέτ, κάτι το οποίο συχνά λέμε στους Κινέζους συνομιλητές μας. Στον συνοθιβετιανό διάλογο υπευλήθη ε, ένα υπόμνημα από πλευράς ε, Θιβέτ ε, για ε, αυξημένη αυτονομία και χαιρόμαστε για το ότι δεν αναζητούν απόσχηση ή ανεξαρτησία και χαιρόμαστε για το ότι ο Δαλάη Λάμα είναι υπέρ της μέσης οδού για να βρεθεί μια βιώσιμη και σταθερή λύση. Χαιρόμαστε για το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ομιλίες, αν και βέβαια δεν υπάρχουν αποτελέσματα ή κάποιος ρυθμός. Οπότε ζητάμε από τις δύο πλευρές να εντείνουν το διάλογο έτσι ώστε να υπάρξει μόνιμη λύση στο Θιβέτ. Από τη δική μας πλευρά μπορώ να σας εγγυηθώ πως εμείς θα υποστηρίξουμε μια τέτοια δικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Εξ τώρα των ομάδων θα λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι. Η κυρία Αντρικιένα για δύο λεπτά. Ο ένατος γύρος συνοθιβετιανών συνομιλιών τελικά δεν καρποφόρησαν και δεν ευελτίωσαν την κατάσταση επιτόπου στο Θιβέτ. Λυπούμεθα γιατί δεν έγινε καμία δήλωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λήξουν οι συνομιλίες και ελπίζουμε ότι τελικά η Ένωση θα εκδώσει δήλωση σχετικά με την αξιολόγηση του πορίσματος των συνομιλιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα ήθελε να ξέρει αν και με ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να συμβάλλει ούτω ώστε να δημιουργηθεί μια αμοιβαίω αποδεκτή λύση για το θηβετιανό ζήτημα ε, και να κατοχυριωθεί η πραγματική αυτονομία για το Θηβέτη και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει για την σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει ήδη ε, την ε, δράση της κοινωνίας των πολιτών στο Θιβέτ αλλά και στις κοινότητες των Θηβετιανών στο Νεπάλ και στο Μπουτάν, των εξόριστων Θηβετιανών για να βελτιωθεί η παιδεία, η πρόσβαση στην αγορά εργασία, τα θέματα ισότητα των δύο φύλων, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η αναβίωση των οικισμών του. Ε, και το σχέδιο της αναβίωσης των καταβλισμών προσφύγων που έχει ε, προετοιμάσει ε, η ε, κοινότητα, η αυτόνομη θηβετιανή κοινότητα θα πρέπει να τύχει της υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχάτως συναντήθηκε στο Λευκό Οικό ο Μπαράκ Ομπάμα με τον Δαλάη Λάμα. Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τον Δαλάη Λάμα στις Βρυξέλλες ούτως ώστε να αρχίσουμε να συντονίσουμε συντονίζουμε τις εθνικές μας θέσεις ε, για το Θιβέτ και να έχουμε μια ομοιόμορφη σαφή ε, ενωσιακή θέση για αυτό το θέμα. Ε, να διορίσουμε έναν ειδικό Ευρωπαίο συντονιστή για το θέμα του Θιβέτ όπως προτείνεται στο νέο πρόγραμμα δράση θα βοηθήσει για να έχουμε προσδιορισμό ενωσιακή θέση και κοινή στρατηγική στο Θιβέτ. Μαρία Μουνίς Δε Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Μουνίς Δε Δύο χρόνια πέρασαν από, τις, από ε, τους ξεσηκωμούς ε, στο Θιβέτ και ελπίζουμε τώρα στην επέτειο να μην ε, επαναληφθούν όλες οι σκηνές βίας που ζήσαμε. Το Κοινοβούλιο τον τελευταίο καιρό εκφράστηκε για την Κίνα και η Κίνα είναι ένας μεγάλος, ε, μια μεγάλη χώρα, είναι ένας πρωταγωνιστής ε, που δεν μπορεί να αγνοηθεί στην παγκόσμια σκηνή. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν η θέση των σοσιαλιστών είναι σαφής. Έχουμε την ίδια θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουμε όμως και το διάλογο, τη σύγκληση και τη συμφωνία. Είμαστε λοιπόν απόλυτα υπέρ της διαπραγμάτευσης ε, και της υπογραφής μιας συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Θιβέτ. Θέλουμε να γίνουν σεβαστά τα θρησκευτικά δικαιώματα στο, Θιβο, στο Θιβέτ, αλλά θέλουμε να έχουμε και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας. Κρίμα που δεν είναι εδώ η αρμόδια επίτροπος, η οποία θα έπρεπε να παρίσταται σε τέτοιου είδους συζητήσεις για εξωτερικής πολιτικής. Και είναι εντελώς άδικο να λέτε ότι η Ισπανική Προεδρία είναι απούς από αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Γκαρίδο είναι συνέχεια εδώ για να, συζητήσει μαζί μας για οτιδήποτε. Η Κομισιόν έχει αρμόδια επίτροπο που θα μπορούσε να είναι παρούσα εδώ και να συζητήσει για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νικόλο Ρινάλντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Φαίνεται σαφές ότι η Κίνα δεν έχει καμία όρεξη να συζητήσει για το Θιβέτε. Η εμπλοκή της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο, οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι συναντήσεις που έγιναν σε επίπεδο ηγεσία στο Πεκίνο δεν οδήγησαν πουθενά. Έχουμε λοιπόν ένα αγώνα μεταξύ Δαβίδ και Γολιάθ με τεράστια δημογραφικά προβλήματα στο Θιβέτ ε, και λήψη δημογραφικών μέτρων που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και καταστολή, βίαιη καταστολή που ζήσαμε πριν από δύο χρόνια. Το, Θιβέ, το Θιβέτ αποτελεί η κληρονομιά της, ανθρω, της ανθρωπότητας, η πνευματικότητά του η μυστικότητά του, η γαλήνη, είναι κάτι τα οποία είναι ακατανόητα για την κινέζικη κομμουνιστική εξουσία. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτιστική γενοκτονία στο Θιβέτ. Εμείς λοιπόν ζητούμε από τους Κινέζους να δεχθούν τον κόσμο του Θιβέτ ε, το Θιβέτ με τις ιδιομορφίες του. Δέχτηκαν λοιπόν μια Κίνα με, το Χονγκ με δύο δηλαδή μέτρα και σταθμά, ας δεχτούν μία Κίνα με τρία μέτρα και σταθμά, δεχόμενη το Θιβέτ όπως είναι. Και αυτό που, που υποσχέθηκε η κυρία Άστον για τον Ευρωπαίο συντονιστή για το Θιβέτ, να μην το ξεχάσει. Πρόκειται για έναν αγώνα ελευθερίας που αφορά στην ταυτότητα της, της Υπήρου μας όταν εμείς θα άρουμε το εμπάργο στα όπλα της Κίνας τότε θα πρέπει να θυμηθούμε και το Θιβέτ. Η κυρία Χέιντι Χάουταλα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να επικρίνω το ότι η Ισπανική Προεδρία έφυγε. κάθισαν να ακούσουν καν την κυρία Αντρικέινε. τους είπε ότι πρέπει να κάτσει εδώ πέρα το Συμβούλιο και να είναι παρόν και να κάνει κάτι για το Θιβέτ. Και εσείς κύριε Πρόεδρε είπατε πως μας είχε προειδοποιήσει η Ισπανική Προεδρία. Ψέμα. Πριν μας είπαν ότι έπρεπε να φύγουν στις 5 αντί για τις 6 παρα 10, αλλά έμειναν για να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία των πολιτών. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό και υποθέτω πως η Κομισιόν είναι σοβαρή και θα κάνει αυτό το οποίο μόλις μας είπε, ότι έχουμε δηλαδή τόσο σημαντική σχέση με την Κίνα που θα πρέπει να μπορούμε να συζητάμε και δύσκολα θέματα όπως το Θιβέτ. Και θεωρώ πως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσουμε την στήριξή μας στο Θιβέτ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Εννέα γύρι διαπραγματεύσεων μεταξύ Κίνας και εξόριστης κυβέρνησης του Θιβέτ δεν είχαν αποτέλεσμα και συμφωνώ με τους συναδέλφους. Φαίνεται πως η Κίνα δεν θέλει αποτελέσματα. Θέλει να συνεχίσει να καταπιέζει το Θιβέτ. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια τέτοια πολιτιστική, πολιτισμική με συγχωρείτε γενοκτονία. Τον προηγούμενο μήνα ήμουνα στην Μαρασάλα, στην Ινδία και συνάντησα τον Δαλάη Λάμα το μίλησα μία ώρα πριν πάει να βρει τον πρόεδρο τον Ομπάμα και ήμουν πεπισμένη πως έπρεπε να σας πω την άποψή του εδώ πέρα. Είναι πολύ πράος άνθρωπος ο Δαλάη Λάμα και είναι κρίμα αυτό το οποίο επιμένει, Κίνα ότι, επιμένει να λέει η Κίνα ότι προκαλεί αναταραχές τις αναταραχές που είδαμε πριν από δύο χρόνια. Αντιθέτως ο Δαλάη Λάμα είπε πως οι Κινέζοι πρόσωποι βεβαίως μπορούν να συναντηθούν με την ε, εξόριστη κυβέρνησή του και αν δείτε τα αρχεία θα βεβαιωθείτε πως δεν προκαλεί αυτό στη βία και όμως αυτό επανέρχεται συνεχώς πρέπει να το καταδικάσει αυτό ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός εάν δεν έχει ε, αν δεν έχει το, θρά, θάρρος η Ευρωπαϊκή Ένωση να στο Θιβέτ το κάνει κανένας άλλος και πρέπει να συγχαρούμε τον πρόεδρο τον ΙΠΑ που τόλμησε να συναντήσει τον κύριο Ομπάμα. Ελπίζω να το κάνει και η ΙΠΑ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κρατήσουμε αυτό το ζήτημα στην επικαιρότητα. Και είπαμε πώ χρειαζόμαστε ειδικό εκπρόσωπο. Έχουμε τόσου ειδικού εκπροσώπου, γιατί δεν έχουμε και ένα ειδικό απεσταλμένο για το Θιβέτ. Έχουμε και προπολογισμό προβλέψει. Ε, αλλά δεν είναι δυνατόν να σηκώνεται και να φεύγει το Συμβούλιο από εδώ μέσα. Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Χάουτ, αλλά... και ένα λεπτό. Ο λαός ε, του Θιβέτ και η βουδιστική κουλτούρα τους είναι ζωντανά στη μνήμη όλων όσων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τότε οι κομμουνιστικές ε, ε, δυνάμεις εισέβαλαν στο Θιβέτ πριν από 61 χρόνια. Οδηγηθήκαμε σε καταστολή τη καθημερινή των Θιβετιανών και στην Λάσα η καταστολή όλων των εξεγέσεων χειροτέρευσε την κατάσταση στο Θιβέτ. Στο μεταξύ από την Ινδία συνεχίζει ο Δαλαϊλά με την ελληνική εκστρατεία του για να βοηθήσει ε, τον ε, Θιβετιανό λαό. Ε, και Ε, το Θιβέτ θα πρέπει να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και αυτό γίνεται βάσει του μάντρα μια χώρα δύο συστήματα που ισχύει στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο. Γιατί όχι στο Θιβέτ λοιπόν. Το Πεκίνο σίγουρα θα μας πει ότι δεν επιθυμείται τέτοια εισβολή σε εσωτερικές υποθέσεις του από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν θετικό και για την εσωτερική πολιτική της Κίνας και για την εξωτερική εικόνα της χώρας στον κόσμο. Ε, θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι και εγώ γιατί δεν εκπροσωπείται η Ισπανική Προεδρία ούτε το Συμβούλιο ούτε η Πατή Εκπρόσωπος ε, το, για την εξωτερική δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ρώση. Μα πραγματικά ε, τα έχω χαμένα. Τα έχω χάσει δηλαδή με, με όσα μας είπε ο Επίτροπος. Εμείς Τι κάνουμε, αναγνωρίζουμε την ε, εδαφική αικαιρότητα της Κίνας, δηλαδή τι εννοούμε. Εννοούμε ότι έχει δικαίωμα η Κίνα να κατέχει το Θιβέτ. Μα και ο Δαλάη Λάμα μίλησε για αυτονομία ε, ε, του Θιβέτ από την Κίνα με στόχο την προφύλαξη της θηβετιανής κουλτούρας και τη διατήρησή της. Πρέπει λοιπόν να σταλεί μία αποστολή επί πού όπως έκανε και ο ΙΕ και να δούμε από κοντά τι γίνεται, να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συντονισμού υποστήριξης του Θηβετιανού λαού που χωρίς την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας θα εκμηδενιστεί. Ο κύριος Μακμίλαν Σκότ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Θιβέτ είναι μια όμορφη χώρα. Ο λαός του είναι ευσεβής, υπομονετικός και καταπιέζεται. Ίσως είναι ο λαός που καταπιέζεται περισσότερο από τους Κινέζους σε αυτή την περιοχή. Και νομίζω πως η επόψηνή μας συζήτηση καταδείξε πως υπάρχει εδώ πέρα συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον οριστή οριστεί π.χ. ένας ειδικός συντονιστής για το Φιβέτα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα γεγονότα μας οθούν να λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Η Κίνα, με συγχωρείτε, ο Google εγκατέλειψε την Κίνα. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα ανθρώπινα δικαιωμάτων εξαφάνιση του Γκάζι Σέγκ, χριστιανού δικηγόρου ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάρος και προσοχή στην Κίνα και στο Θιβέτ και να συμπενθυμίσω πως με την παγκόσμια έκθεση της Αγκάης που ανοίγει τον Μάιο όλοι όσοι επιχειρούν στην Κίνα πρέπει να σκεφτούν το σύμφωνο του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις. Τέλος, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ορίσει ειδικό απεσταλμένο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ορίσει έναν εισηγητή για το Θιβέτ. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα, συνάδελφοι, στους ομιλητές που έχουν καταγραφεί. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κατσμάρεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ το θέμα του Θιβέτ ε, δυστυχώς είναι σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι τόσο άσχημο όσο πριν από δύο χρόνια, όσο όταν είχαμε εξεγέρσεις, επεισόδια, δολοφονίες, αλλά ακόμα και τώρα συλλαμβάνονται μαθητές που προσπάθησαν να τιμήσουν την επέτειο αυτή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον πολιτισμό της περιοχής τους οι κινέζικες αρχές θεωρούν ότι ο Δαλάη Λάμα είναι κάποιος ιδιώτης. Έτσι ακριβώς λέγανε και το Λεχ Βαλέσα οι κομμουνιστές πριν από 25 χρόνια. Νομίζω πως ε, και ελπίζω να έχει ανάλογη κατάληξη και αυτή η υπόθεση. Σήμερα δε στην Ταραμψάλα έχουμε την 21η συνεδρίαση της λεγόμενης task force ε, για το Θιβέτ, ε, δηλαδή ενός ε, σύνοθιβετιανού διαλόγου και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει σε αυτόν τον διάλογο. Πρέπει όμως να είναι μια πραγματική συζήτηση. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε κάτι και είναι λυπηρό το ότι δεν είναι παρόν το Συμβούλιο γιατί στο Συμβούλιο απευθυνόμαστε. Το Συμβούλιο στέλνει ειδικού απεσταλμένους και το τονίζω γιατί ζητήσαμε και στα ψηφίσματά μας ε, ειδικό αποσταλμένο για να μπορέσουμε να ασκήσουμε κάποια επιρροή για να έχουμε συνομιλίες μεταξύ Θιβέτ και Κίνας και κάτι ακόμα δεν αντιλαμβάνομαι το ότι το 2004 διοργανώνει πάλι Ολυμπιακούς Αγώνες Ολυμπιακούς Αγώνες Νεολαίας η Κίνα και δεν υπάρχει καμία πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λυπηρό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μπαϊσδί για 1,5 λεπτό. Meggyőződésem, hogy leegyszerűsített képünk van a tibeti folyamatokról. Ott egyszerre... Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αφενό υπάρχει ένα εξυγχρονισμό στη χώρα, από την άλλη δικαίωση υπάρχει κάποια κριτική. Πράγματι νομίζω πως ε, μία διευρυμένη και πραγματική αυτονομία θα προσφέρει λύσεις. Το δε Πεκίνο νομίζω αναφέρθηκε το ότι μπορεί να υπάρξει μία χώρα δύο κοινωνίες και εδώ πέρα μπορεί να υπάρξει μία χώρα δύο θρησκείες. Δεν είναι τόσο δύσκολο Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σε αυτά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ρωμάνεο ο Πρόντι, η κυρία Φέρε, ο Βάλνερ, η Μάρκοτ Βάλστρομ είναι άτομα που χαίρουν εκτίμησης. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Και η κυρία Άστον πρέπει, έπρεπε να είναι παρούσα. Μιλάμε πάρα πολύ για τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνας. Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβουλίο δεν το έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα, ποτέ. Στις δε ε, συζητήσεις για σχέση με την Κίνα, ποτέ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εμείς ε, επιτυχεί σε αυτό. Λίχτεμπεργκ απουσιάζει, οπότε τσαρνέκι ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε διότι διεξάγεται αυτή η τόσο σημαντική συζήτηση με τόσο λιγάριθμους παρισταμένους. Η κυρία Άστον θα έπρεπε να είναι εδώ. Ε, δεν θα πρέπει να πηγαίνει μόνο στα, στις πολύκροτες εκδηλώσεις Όπω εχθές, παραδείγματο χάρη, παρουσίασε το πρόγραμμά τη για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Είναι σημαντικότατη η πρόκληση και πρέπει να ακούσουμε την άποψή τη, είτε είναι θετική είτε αρνητική. Θα έπρεπε να είναι εδώ η κυρία Άστον. Και δηλαδή την ύβη σχήρα τη. Ε, έτσι μου φαίνεται πολλές ε, πολλά κράτη που ε, εκπροσωπούνται εδώ επιθυμούν να έχουν ε, εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα και ξέρω πόσο δυσάρεστο είναι να κατακρίνει κανείς την Κίνα. Αλλά δεν μπορεί να ανήκει έτσι τα σχήρες κυρία Άστον. Ευχαριστώ Μέλτσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούμε τελευταία για πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις ε, και φυλακίσεις όταν ε, βεβαίως ε, ανέλαβαν οι κοινές τη του Θιβέτ μιλούσαν για απελευθέρωση των Ιμαλαίων κάτι το οποίο βεβαίως πλέον έχει ακουστεί ηρωνικό και βεβαίως εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία παράνοια με αυτή που έχουν επιβάλει στο Αφγανιστάν και το Ιράκ οι οποίες παρόλα αυτά υποστηρίχθηκαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και βεβαίως ε, πρέπει να γίνει σεβαστός και ο πολιτισμός τους και όχι να γίνει μόνο folklore για τους τουρίστες. Και μάλιστα είχε δηλώσει η Κίνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 πως είναι διατεθειμένη για συνομιλίες, αλλά τίποτα δεν έγινε. Πρέντα μετά για δύο λεπτά. Ο κύριος Κατσμάρεκ αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες του 2008. Πέρασαν δύο χρόνια και δεν ξέρουμε πόσοι κρατήθηκαν ή κρατούνται. Δεν ξέρουμε πόσοι απολευθερώθηκαν. Εκείνο όμως που ξέρουμε είναι ότι όλοι αυτοί διαδήλωναν ειρηνικά ανεμίζοντας τη θηβετιανή σημαία και μοιράζοντας προκηρύξεις. Περάσανε λοιπόν δύο χρόνια και δεν έχουμε ιδέα πότε συνελήφθησαν και τιμωρήθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. η παρεμβατικότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος στα του Θιβέτα πετώντα γρήγορες δίκες και παραδειγματικές ποινές είναι κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Πρέπει λοιπόν και το υπογραμμίζω να έχει η Ευρώπη μία κοινή θέση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται άμα δεν έχουμε μία κοινή θέση. Οι κομμουνιστές προσπαθούν να εκφοβήσουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης ένα προς ένα. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα μέσο ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. Πρέπει να λυθεί σε επίπεδο διάσκεψης κορυφής. Η κυρία Άστον που συναντήσαμε χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αναγνώρισε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη θέση μας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει δίκιο. Ευχαριστώ Μιγκάλσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια ε, ε, επιχείρηση μπορεί να κερδίσει, κερδίζει χρήματα εις βάρος ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς μπορεί να συμπεριφέρονται έτσι οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δεν υπερασπιζόμαστε αυτές τις αποκαλούμενες ευρωπαϊκές αξίες. Ε, θα έπρεπε να είναι εδώ η κυρία Άστον για να ακούσει αυτές τις απόψεις. Και αποχωρούν από την αίθουσα εκπρόσωποι του Συμβουλίου με το που αρχίζει η συζήτηση για το Θιβέτ. Ο αγαπητός κύριος Επίτροπος μας είπε ότι υπάρχει ένας διάλογος και νομίζω ότι αστιεύεται η κινέζικη κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να αρχίσει το διάλογο. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά, ο κύριος Κελ. Η κληρονομιά, η πολιτιστική του Θιβέτ είναι η κοινή μας κληρονομιά, είναι προς το κοινό μας συμφέρον, η ταυτότητα, η θρησκεία και η γλώσσα του να διατηρηθούν και να απτυχθούν με τις καλύτερες συνθήκες. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει υπό το κάλυμα της βιομηχανικής ανάπτυξης υπάρχει πολιτισμική γενοκτονία. Και οι Φιβετιανοί πάνε να γίνουν μειονότητα στη χώρα τους. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μόνο με το να αποκτήσουν ουσιαστική αυτονομία με έναν διάλογο επικοδομητικό χωρί προκαταλήψεις το ασύλλητο και τι δύο πλευρέ. Δεν έχω αμφιβολία, κύριε Επιτροπέ, που... για αυτό το οποίο δηλώνεται πω ανισχύεται πραγματικά για το Θιβέτ. Ως αποτέλεσμα ενός τέτοιου διαλόγου και με το να ανοίξει το Θιβέτ για τα ξένα μίμιε και ειδικού ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει να κερδίσει τα πάντα η κινέζικη κυβέρνηση και κυρίω διεθνώ Η Κίνα θα γίνει πραγματικά μεγάλη μόνο εάν σεβαστεί τις μειονότητες. Ως χειρονομία καλής θέλησης, ο Δαλάη Λάμα που αναγνωρίζεται παγκοσμίω θα πρέπει να μπορέσει να επισκεφτεί την πατρίδα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκμεταλλευτεί την ε, συνθήκη της Λισαβόνας για να αναπτύξει επαφέ με ένα έθνος που απειλείται η ύπαρξή του και το φυσικό του δικαίωμα για αυτονομία και πολιτισμό παραβιάζεται. Υποστηρίζω το ότι η κυρία Άστον πρέπει να συναντήσει τον Δαλάη Λάμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει ειδικό εκπρόσωπο για το Θιβέτ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ Στάσνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, 10. marca sme si pripomenuli... Εορτάσαμε ε, την ε, ε, επέτειο και της ε, κινέζικης εισβολής στο Θιβέτε και των εξεγέρεσεων στη Λάσα ε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το ότι η Κίνα προσπαθεί να αφομοιώσει το, τους Θηβετιανούς και να εκμηδενήσει ε, τον πολιτισμό τους. Όλοι ξέρουμε γιατί είναι ε, ικανή η Κίνα. Ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Ασίας που χρονολογείται εδώ και χίλιοι κινδυνεύει να εκλείψει. Δεν μπορούμε να μείνουμε άπρακτοι. Υπάρχει ομάδα των φίλων του Θιβέτ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίστοιχε ε, ομάδε υπάρχουν άνα τον κόσμο, στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ, στην Ινδία, γενικότερα στην Ασία, στη Σλοβακία θα συσταθεί μια τέτοια ομάδα φίλων του Θιβέτ και νομίζω ότι εάν διαμεσολαβήσουμε στι ε, διαπραγματεύσει που γίνονται ανάμεσα στι Κινέζικε Αρχέ ε, και το Δαλαϊλάμα μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα και των Θιβετιανών προσφύγων που ε, ζουν ε, ε, υποχείριστες συνθήκες σε γειτονικέ χώρες. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ξεχνά αυτούς τους πρόσφυγες. Ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Κάτσε διάι. Το Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η συζήτηση αυτή μας ικανοποιεί γιατί φαίνεται πως συμφωνούμε αλλά όλο τέτοιες συζητήσεις κάνουμε και είμαστε έτσι φιλάνθρωποι αλλά τι είμαστε τελικά υποκριτές και εγώ το ίδιο και εγώ κινέζικα αγαθά αγοράζω και όλοι μας Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε σαφώς κατά αυτών των καταστάσεων και ένα πρώτο σημαντικό βήμα είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε σήμερα ήδη. Δηλαδή, ο ορισμός ενός ειδικού απεσταλμένου για το Θιβέτ. Κάποιος ο οποίος θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις εξ ονόματός μας. Για να μπορούμε να πούμε τελικά πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια αξία στην οποία δεν συμβαζόμαστε. Το να μιλάει κανείς εδώ και σήμερα για το Θιβέτ είναι θέμα δικαιοσύνης και ευθύνης. Λοιπόν, κρίμα για αυτούς που πίστευαν ότι δεν θα έπρεπε να το συζητήσουμε. Χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και λυπούμε να διαπιστώνω ότι παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει ε, ο Δαλαϊλάμα για να έρθει σε επαφή με, τον, με τις κινέζικες ε, αρχές συνεχώς τροχοπεδείται από τις αρχές αυτές. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε ούτε να τροφοδοτούμε αυτή τη στάση ούτε να βοηθάμε την Κίνα ή να κοιτάμε σαν απλοί παρατηρητές. Πρέπει εμείς να, μιλά, να, να το έχουμε καθαρά στο κεφάλι μας ότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν λύση στο πρόβλημα είναι η Κίνα και είναι δεσμευμένη η Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, θα πρέπει να δεχθεί η Κίνα ότι θα υπάρχει ένα οικονομικό κόστος όταν δεν τα δέχεται όλα αυτά. Αλλιώς ποτέ δεν θα είμαστε αξιόπιστοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, Τούκους. Chairwoman, Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες μέρες ε, τιμήσαμε την 51η επέτειο της εξέγερσης του Θιβέτ. Έκτοτε ο Δαλάη Λάμα προσπαθεί να εκπροσωπήσει τον λαό του και προσφέρει ένα υπόδειγμα στον κόσμο για το πώς μπορεί κανείς να επιδιώξει δημοκρατία χωρίς βία. Οι Ευρωπαίοι διδάσκονται από τον Παναγιώτατο. Πρόσφατα εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τους Ουιγούρους, τη μειονότητα αυτή, και με την Αουνξάν Σουνκή και άλλους ε, δημοκράτες ε, αντιφρονούντες και εδώ πέρα βεβαίως είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και εγώ ως Ούγγρος μειονοτικός της Ρουμανίας σας ευχαριστώ όμως ακολουθεί ο κύριος Ομπερμαϊερ λέει η πρόεδρος. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Επίτροπο. Για εμένα το Θιβέτ είναι μια χώρα υποκατοχή και νομίζω πως πάρα πολλοί σε όλες τις ομάδες εδώ πέρα τις κοινοβουλευτικές συμφωνούν ε, μαζί μου. Νομίζω υπάρχει και η σχετική συνάντηση με την Κίνα το φθινόπωρο πρέπει να τεθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς βεβαίως γρήγορα καταδικάζει κάτι μικρές ε, χώρες ε, εκεί πέρα που δεν έχουν και καμία ισχύ. Αλλά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για μεγάλες και σημαντικές χώρες, οικονομικά σημαντικές χώρες. Εκεί πέρα είμαστε πολύ πιο διπλωμάτες. Δεν είναι... Ε, πρέπει επιτέλους να επιτύξουμε και λίγο ανάστημα και λίγη ραχοκοκαλιά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πιέσουμε και με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αναμένω τοποθέτηση από την είπατε εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ. κατόπιν. με τις μου είπε πριν κρατκιμ δάνα Εγώ πριν από λίγο καιρό κατάφερα να πάω στο Θιβέτ. Γίνονται πρόοδοι Πρόοδοι όμως οι οποίες είναι ε, προς την αρνητική κατεύθυνση και όχι προς τη θετική, δηλαδή περιθωριοποιούνται οι παραδοσιακές πνευματικές αξίες, περιθωριοποιείται η παραδοσιακή φιβετιανή ε, ευνοείται μία σύγχρονη εικόνα, μια μοντέρνα εικόνα του Θιβέτ, μολύνονται τα ποτάμια, ε, παραμορφώνεται το τοπίο από αυτοκινητοδρόμους. Ζητούμε λοιπόν οι προσδοκίες μας από την Κίνα να είναι αρμονικές με την πραγματικότητα ούτως ώστε το Θιβέτ να μην γίνει μουσείο αλλά χωρίς να καταστρέφεται. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Κάτσε, διάκομαι ε, τον Επίτροπο τώρα, κύριο Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, από τη σημερινή συζήτηση ότι ανησυχούμε πραγματικά για την κατάσταση στο Θιβέτ και επισημάνθηκε ε, στις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι είναι θεμητές αυτές οι ανησυχίες. Έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από την ε, ε, εισβολή της Κίνας στο Θιβέτ από το 1959 και πρέπει ταχύτατα να επαναληφθεί ο διάλογος ανάμεσα στα δύο μέρη, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Ε, ορίζουμε την ε, πανεκκίνηση του διαλόγου το Σεπτέμβριο του 2009 ανάμεσα στο Δαλαϊλάμα και τις Κινέζικες Αρχές. Ελπίζουμε να καρποφορήσει ο διάλογος, να έχουμε θετικά αποτελέσματα και να δοθούν λύσεις, βιώσιμες λύσεις για το Θιβέτ. Ε, στον ε, πολιτικό διάλογο και στις περαιτέρω επαφές με την Κίνα, ε, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ε, κινέζικες αρχές να ρυθμίσουν όλα τα εκρεμή ζητήματα σε σχέση με το Θιβέτ. Η Κίνα θεωρεί βέβαια ότι είναι εσωτερικό ε, το θέμα, θέμα εσωτερικής πολιτικής ε, και ενημερώνει συστηματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άποψή της για αυτό το θέμα. Δεύτερον, τονίζω ότι υπάρχει και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου με την Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά τονίζει πόση σημασία αποδίδει στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης ε, στο Θιβέτ. Ε, παρακολουθούμε εκ του σύναγκης ε, την πορεία των ε, συνομιλιών και συνεχίζουμε τις επαφές με τον Δαλαϊλάμα και τους εκπροσώπους του. Την, τον περασμένο μήνα ενημερωθήκαμε για τον έσχατο γύρο συνομιλιών και από τα δύο μέρη και τους ενθαρρύναμε και πάλι να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο. Κλείνοντας, ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω ότι ε, βλέπω την συνεχή δέσμευση και αφοσίωση του Κοινοβουλίου για να προαχθεί ο πολιτικός διάλογος ε, για το Θιβέτ. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ως προς την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των προσωπικών δικαιωμάτων στο Θιβέτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγη εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αξιότιμοι συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο